29 υπέρ, 23 κατά. Α, γίνεται δεκτή επομένω. 9. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, εκπίπτει. 14 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα εκπίπτει, δεύτερο εκπίπτει, το τρίτο όμως μπορεί να ψηφιστεί. Ψήφι υπέρ του τρίτου τμήματος στις 14, υπέρ. Κατά. Απόχες, εγκρίνεται. 15, υπέρ. Κατά. Απόχες, δεκτό. 19, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 16 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεκτή ήμουν. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 22 υπέρ. κατά αποχές δεκτή 23 εκπίπτει όχι όχι ψηφίζεται υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 23 παρακαλώ πάμε ψηφίσατε όλοι πέρας 27-21 με 6 αποχές γίνεται δεκτή. 23 πάμε. Στην 24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές <clears throat> απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή εκπίπτει λοιπόν η 30 πάμε στην 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 εκπίπτει 33. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονικά για τη 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 35 υπέρ, 20 κατά, σαφώς εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 40 υπέρ. Πέτερ. Είχα ζητήσει από τη γραμματεία και στο είχα ζητήσει από τον εισηγητή και το σκιώδη εισηγητές να γίνει μια προφορική τροπολογία κάπως ε, διευκρινίσαμε τη γλωσσική μορφή για το αγγλικό κείμενο και προτείνω το εξής. Πρόκειται για τη χρήση προϊόντων από ζώα. Το αρχικό κείμενο της κυρίας Λιωτάρτ αφορούσε μια απόλυτη απαγόρευση για την επόμενη γενιά σε περίπτωση προβλημάτων σε μια αγέλη ζώων. Αλλά εμείς θέλουμε να περιορίσουμε λιγάκι αυτή την απόλυτη απαγόρευση Γι' αυτό θα πρότεινα μια τροποποίηση στο κείμενο της ισίδης, που λέει μια νομοθετική πρόταση η οποία αφορά την απαγόρευση κλωνοποίησης και εμπορίας προϊόντων από κλωνοποίηση καθώς και μια κανονιστική ρύθμιση για τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από την επόμενη γενιά. <clears throat> Αυτό επανέρχεται στην θέση που είχε εγκρίνει στο παρελθόν η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε να εγκρίνουμε αυτή την τροποποίηση είτε στο σημείο 3 είτε στο τελευταίο σημείο. Μπορεί να τεθεί αυτή η πρόσθετη φράση. Να ψηφίσουμε καταρχήν την προφορική τροποποίηση του Πέτερ Λίζερ είναι η προφορική τροπολογία υπαριθμών 2. Είναι σωστό αυτό. Έχουμε το ίδιο κείμενο. Λοιπόν, πρώτα τη 40 της ε, Julie Gerling και μετά την προφορική τροποποίηση του Πέτερ Λίζ. Εντάξει. Τροπολογία 40 Gerling υπέρ <coughs> κατά αποχές απερίφθη. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα η τροπολογία υπαριθμών 2 του Πέτερ Λίζε ψήφι υπέρ Συγγνώμη, μήπως μπορεί να ξαναπεί ο κύριος Λίζε πού θα βάλει την προφορική του τροπολογία. Ψηφίζουμε την 2, όπως αναφέρεται στο κατάλογο ψηφοφορίας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Λίζε να μας εξηγήσει τι ακριβώς λέει το κείμενο. Ναι, ναι, βεβαίως. Στην Παύλα 3, στο αρχικό κείμενο της κυρίας Λιωτάτ, περιλαμβάνει μια απαγόρευση της κλωνοποίησης και την εμπορία προϊόντων από την επόμενη γενιά. Εμείς όμως στο παρελθόν είχαμε μια θέση ως κοινοβούλιο όπου είχαμε ζητήσει όχι μια απαγόρευση για τη χρήση προϊόντων από την επόμενη γενιά κλωνοποίησης, αλλά να υπάρξει μια ρύθμιση στα θέματα αυτά. Και επομένω υπάρχει αυτή η προφορική τροποποίηση που λέει ότι θα υπάρξει μια νομοθετική πρόταση που να εφαρμόζει μια ε, απαγόρευση κλωνοποίησης και εμπορίας προϊόντων κλωνοποίησης και επίσης ένα κανονισμό για τα, την επόμενη γενιά και τα προϊόντα από την επόμενη γενιά. Αυτό θα αντικαθιστούσε λοιπόν στο εδάφιο 3 το αρχικό κείμενο της κυρίας Λιωτάτ. Για να είμαστε σαφείς. Είναι η τρίτη παύλα, τρίτο εδάφιο του 4, του αρχικού κειμένου της κυρίας Λιωτάρτ. Αυτό το οποίο σας ανέγνωσε ο Πέτερ Λίζε. Και αυτό θα ψηφίσουμε τώρα. Ωραία. Η συγκίτρια τώρα έχει το λόγο. Ε, Ειλικρινά πιστεύω ότι εδώ είναι ζωτική σημασία θέματα αυτά και μια προφορική τροπολογία εγώ δεν θα την ήθελα, δεν θα ήθελα προφορική τροπολογία σε αυτά τα θέματα. Συνεπώ δεν ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. Δεν θα ψηφίσουμε λοιπόν και κάναμε χωρίς ε, λόγω όλη αυτή τη φασαρία. Περνάμε στην τροπολογία 43, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προφορική τροπολογία 1. Για την 44 υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Μπορούμε λοιπόν να την ψηφίσουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 έλεγχος ηλεκτρονικός. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 32 υπέρ 25 κατά εγκρίνεται. Σαράντα υπέρ. 47 συγγνώμη κατά. Αποχές. Και πάλι. Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην ψηφοφορία. 47 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή με μικρή διαφορά 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα ψήφισατε όλοι πέρας 34-19. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικά ελέγχουμε για την 53. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 27-20 γίνεται δεκτή. Με 11 52 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 54 εκπίπτει, 56 ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή, 58 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται, 57 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται, 60 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ 67 λοιπόν είπαμε πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας 26-30 απορρίπτεται. 69. Υπέρ. Κατά. Απόχες, εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Ασαφέστατη η κατάσταση. Ηλεκτρονικά για την 74. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 26-25. Έπρεπε να ψηφίσω όχι, λέει ένας, ο Καλ Σλούτερ. Είναι πολύ εύκολο να διαλέξετε το σωστό. 26-25. Λοιπόν, γίνεται στο τσίμα τσίμα δεκτή. 64 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ. Υπέρ, υπέρ για την 64. Υπέρ. Κατά. Απόχες Απορρίζεται. Έλεγχος για την 64 ηλεκτρονικός. Ο κύριος Λίτερ θα πρέπει να ψηφίσει σωστά. Ψηφίσατε όλοι περασε 29 29-28. Μπράβο Καλ Σφίτερ, μπράβο. Εβδομήντα εννέα Αρσένης υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 80 υπέρ. Κατά. Έλεγχος ε, για την 80. Ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της οφορίας. 60. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. 81 υπέρ. Κατά. αποχέ δεκτή. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή 77 υπέρ κατά εγκρίνεται και τώρα η τελική ψηφοφορία για το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Καρλ και εσύ. Πέρασε προφορίες. 33 υπέρ 16 κατά 11 αποχές. Γίνεται δεκτή λοιπόν η γνωμοδότηση συγχαρητήρια στην κυρία Λεωτάρντ. Τώρα περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Πρόκειται η τροποποίηση κανονισμού 1760-2000 σχετικά με την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοηδών και την κατάργηση των διατάξεων σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βοηού κρέατος. Η κυρία Σοφία Κονή είναι η συγκήτρια. Ψηφίζουμε λοιπόν, αλλά δεν θα παρακολουθήσουμε ακριβώς το κατάλογο για το 59 και το 62 της κυρίας ε, Μπέρεντ. Θα ψηφιστούν ε, χωριστά. Πρόκειται για τα άρθρα 11 και 1. Συνεπώς, Συνεπώς, αρχίζουμε με την οδηγία. Η μικρή ψηφοφορία πρώτα. Τρία. Τροπολογία αριθμός 3. Ψηφίζουμε. Ξεκινάμε με την οδηγία, έτσι, επειδή η οδηγία είναι πιο σύντομη, λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία αριθμός 3. Μπαρτ Στάς, Λιωτάρ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία αριθμός 1. Δεν κρίνεται. 4 και 5 τώρα. Καταπίπτουν. Τροπολογία 1. Άγκρι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 έχει αποσυρθεί. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα ψηφίζουμε, τελική ψηφοφορία. Εντάξει, ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 59 ψήφοι υπέρ. Καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται συνεπώς Τώρα, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε και το κείμενο νομοθετικού περιεχομένου. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορία. 60 υπέρ, καμία ψήφος κατά, ούτε αποχές. Ωραία. Περνάμε τώρα στην ε, πιο μεγάλη μας ψηφοφορία και αρχίζουμε με το C1. Υπέρ, παρακαλώ. Είναι συγκεντρωμένες ψηφοφορίες αυτές. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σε δύο υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το C2. Ψηφίσατε όλοι. Κάρλ Σούλτερ, ψήφισες όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 33 ψήφοι υπέρ εγκρίνεται. Σε 3 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία πάλι. Σε τρία λοιπόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 37-23 το αποτέλεσμα εγκρίνεται. Σε 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σε πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σε 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, Ψηφίζουμε για την τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α, όχι, απορρίπτεται, απορρίπτεται. Σε 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, σε ελέγξουμε παρακαλώ. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για την 56. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 32 κατά, απορρίπτεται. Άγκρι 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. «58 έχει απορριφθεί». Μα το είπαμε ότι θα απομακρυνθούμε από τον κατάλογο που έχετε μπροστά σας. όσον αφορά τις τροπολογίες Νέλχαρτ και Ροτμπέρε. Τώρα 59. Ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Και ο Καρλ Σούλτερ. Άρα μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. 18 υπέρ, 41 ψήφι κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εξιδενα κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, κατά πίπτη. Και πρέπει άρα να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα μόνο. Στα γαλλικά από τη μετάφραση δεν έχω όλο όλη τη μετάφραση δεν καταλαβαίνω αν έχει περάσει δεν έχει περάσει. Ας πούμε για την τροπολογία 5 δεν κατάλαβα το πρώτο τμήμα πέρασε, απορρίφθηκε, τι έγινε. Zu 5, Frau Kollegin, sind beide Teile angenommen. 5 και τα δύο τμήματα έχουν εγκριθεί στην 5. 61. Δεύτερο τμήμα. Εκεί μόνο το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε στην 61. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. 62 λοιπόν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 62. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίες. 23 υπέρ, 37 κατά. Απόρριπτεται. Άγκρι 11 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 75 λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 77 και 78 μαζί για την ίδιες. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Άγκρι 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 17 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άγκρι 17. Ψηφίστε παρακαλώ, πέρα στις φοφορίες. 36 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται. Τώρα 79 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Για να ελέγξουμε παρακαλώ την 70. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορίες. 36 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται. Η 71 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ και 78 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 17 Α, όχι, 18. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 80. Τροπολογία 80. Λοιπόν, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Η 26-29 και μια αποχή. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. 82. Θα ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. 28 υπέρ, 31 ψηφί κατά. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε και εδώ ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την 81. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις 47 υπέρ 12 κατά εγκρίνεται. Σηκώνετε καλά τα χέρια παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος, για να μπορούμε να ψηφίσουμε. Τα τρία. Υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικά. 83. Ηλεκτρονικά ελέγχουμε παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορίες. 28 υπέρ, 31 ψήφι κατά, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 85 86 87, 88, 89, 90, 91 92 και 93. Μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Επαληθεύουμε λοιπόν την ψηφοφορία για όλες αυτές τις τροπολογίες μαζί. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 34 υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνονται οι τροπολογίες αυτές. 98 steht da. 98 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 καταπίπτει. 100 επίσης. 101 επίσης. 102 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104. Υπέρ. Κατά. 104 ήμασταν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105 καταπίπτει. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις τώρα. Ρυθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12, 13 και άγκρι 2 και 14. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις φοφορίες. 40 υπέρ, 18 κατά. Μία αποχή. Εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, α, μια στιγμή. 21 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Α, στη 19. Πρέπει να ελέγξουμε για τη 19. Συφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. 24 τώρα. Είπαμε κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Α, όχι. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Έτσι θα έλεγα εγώ. Θα ελέγξουμε. Εντάξει. Ψηφίστε λοιπόν για την 27. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη 25 υπέρ, 34 κατά. Καμία αποχή. Απορρίπτεται. 28 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 40. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ας ελέγξουμε παρακαλώ για την ε, 41. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις φοφορίες. Απορρίπτεται. 26 υπέρ, 32 κατά. 42 και 44 καταπίπτουν. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 45. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τελευταία αυτή τροπολογία. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 30 υπέρ, 28 κατά. 45 εγκρίνεται λοιπόν. 53 53 Υπέρ. Κατά. Να επαναλάβουμε. Τροπολογία 3 και τροπολογία 53. Μαζί είναι ίδιες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα, περνάμε στην τροποποιημένη ε, γνωμοδότηση. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ψηφίσατε. Πέρα τη ψηφοφορία. 30 ψήφοι υπέρ, 15 κατά και 13 αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα μας μένει το κείμενο νομοθετικού περιεχομένου, πάλι με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 31 ψήφοι, 5, 16 κατά, 12 αποχές. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. 11 σημείο, 11 στην ημερήσια διάταξη παρακαλώ. jetzt kommen wir zu 11. Änderung der Richtlinie 64 432 EWG. Wir stimmen Τροποποίηση της οδηγίας 64-432, συμβιβασμός 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, τρι, τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το 55 μάλλον κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται επίσης. 56 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 60 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 61 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. στο δεύτερο τμήμα, δεν είμαι σίγουρος, ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Α, δεν ψήφισαν ακόμα όλοι. 30 ψήφοι υπέρ 25 κατά, επομένως εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο 74. Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το 77, παρακαλώ. Εψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. 27 υπέρ 27 κατά και επομένως απορρίπτεται. 81. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 82. Υπέρ, κατά, κατά, αποχές απορρίπτεται. 83, 84, 85, 86, 87, 88 αυτά αποσύρονται. 89 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνον, εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν έχουμε αποτέλεσμα. Λοιπόν, 17, 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 96 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για το 96 με προφορική τροπολογία. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. 34 ψήφοι υπέρ, 20 κατά και επομένως εγκρίνεται μία αποχή. Ήτρε 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ ε, ηλεκτρονική επαλήθευση εντάξει ηλεκτρονική επαλήθευση για το 25 άρχεται η ψηφοφορία εψήφισαν όλοι πέρας Απορρίπτεται 23-32. 26 ε, υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση και για το 26 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 28 ψήφοι υπέρ, 26 κατά, επομένως εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που έχουν ψηφίσει δύο φορές. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Εψήφισαν όλοι πέρα της πληροφορίας. 23 ψήφοι υπέρ, 32 κατά, επομένως απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 110α, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Δεύτερο τμήμα λέμε. Α, όχι, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για το δεύτερο τμήμα. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ε, ναι. Συνεχίζουμε με τον κατάλογο ψηφοφορίας. Δε, σελίδα 14. Δεν την έχουμε. Ψηφίζουμε την 35. Ο εισηγητής είναι υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 36 άρχεται. Ψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες, 27 υπέρ 28 κατά, επομένως απορρίπτεται. Απορρίπτεται με διαφορά μιας ψήφου, πάντως απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 8 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38. Όχι, 138 διορθώνει ο Πρόεδρος, 138. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ 143 λέει ο πρόεδρος. 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 45 β υπέρ. Κατά. Προβληματίζεται ο πρόεδρος. Εγκρίνεται πάντως. 46. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 154, ε, α όχι, ηλεκτρονική επαλήθευση για το 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 30 ψήφοι υπέρ, 26 κατά, επομένως, η 47 ενεκρίθη. ενεκρίθη. Περνάμε λοιπόν... 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήτρε 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της Ήτρε 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ήτρε 3 εγκρίνεται. 32 ψήφοι υπέρ, 24 κατά. Ήτρε 4 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση επί της Ήτρε 4, πολύ ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία, εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. 33 ψήφοι υπέρ, 23 ψήφοι κατά. Επομένως είναι σαφές το αποτέλεσμα, εγκρίνεται. 49 και ήτρε 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα του 3. Το πρώτο τμήμα μόνο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50-51 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Είναι ταυτόσιμες. 52-53 ταυτόσιμες υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 1 Α, η ηλεκτρονική επαλήθευση του 52-53 ψήφισαν όλοι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 αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία επί της τροποποιημένης πρότασης, με ηλεκτρονική ψηφοφορία φυσικά, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 49 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, 6 αποχές και επομένως θετικό το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε τώρα επί του νομοθετικού ψηφίσματος η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Και εδώ έχουμε 48 ψήφους υπέρ, μία ψήφο κατά και τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Περνάμε επομένως στο επόμενο σημείο. Ordnungspunkt 13. Το σημείο 13 της τη διάταξης. Τα ύδατα. Με εισηγητή τον κύριο Ρίχαρδο ΖΕΕΔΕΡ Και ξεκινάμε αμέσως. Τροπολογία 24. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το, το 6 θα το ψηφίσουμε. Τροπολογία 1, ε, παγιοποιημένη, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9α υπέρ πετησιό κατά αποχές εγκρίνεται παγιοποιημένοι 2 ενοποιημένοι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 519 19 δεν ψηφίσουμε, 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 516 16 υπέρ κατά Απόχες. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 38 υπέρ. Κατά. Απόχες. 5 Πέτη 12α. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές δεχτεί. Πέτη 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεχτεί. 39. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεκτή. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 40 υπέρ. κατά αποχές δεκτή. Ενοποιημένη 3 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για τη 45 έλεγχος. Για την 95 πρώτα. Εντάξει, 95 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Για την 95 λέει ο πρόεδρος. Όλοι ψηφίσατε. Πέρας. 24 υπέρ, 30 κατά. Από απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 48 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για 48. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 29 υπέρ, 24 κατά. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την 49. Όλοι ψηφίσατε. Πέρας. και όχι εγκρίνεται. 30 με 21. Γίνεται δεκτή. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 18 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 52. Έλεγχος ηλεκτρονικός για την Ήτρε 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. «27 με 25». Γίνεται πράγματι δεκτή 18 Ήτρε. 27-25 λοιπόν είναι δεκτή. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πεν... Έλεγχος στην 52. Μάλιστα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 24-26 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν σαφώς. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ήτρε 20 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 60 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 62 υπέρ, κατά αποχές δεκτή,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 οι φιλελεύθεροι και υπέρ και κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το τρίτο τμήμα της 64. Όλοι ψηφίσατε. Πέρασε. Εγκρίνεται και το τρίτο τμήμα, 27-24. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 79. Θέλουμε έλεγχο βεβαίως. Ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 72. Πάμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα της 72. 79. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Έλεγχος ηλεκτρονικός 79 τμήμα 1. Πάμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 30-25 γίνεται δεκτό. Δεύτερο τμήμα της 79. Ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτό. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές <clears throat> δεκτή. Πέτει υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 14 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνευση. 75 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος το 75 τμήμα 2. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 31 με 20 γίνεται δεκτό το δεύτερο τμήμα. 76 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήτρε 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πέτει 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πέτει 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πέτει 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πέτει 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πέτει 18 υπέρ έλεγχος για την 5-15 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. απορρίπτεται η 15 5 5 18 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ενοποιημένη 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Πάμε στην ήτρα 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ενοποιημένη 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 88 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συ, ενοποιημένη 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. χωρίς μικρόφωνο. Ναι, ναι, ψηφίσαμε. Ναι, ναι, όλα είναι εντάξει, όλα βαίνουν καλώς. Ενοποιημένη 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 96. Με προφορική τροποποίηση. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ήτρε 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 107 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ήτρε 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 104 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 106 σε δύο τμήματα. Τμήμα 1 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 111 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 112 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 521 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 512 β. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Ήτρα 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήτρε 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή 115 υπέρ κατά αποχές δεκτή 520 υπέρ κατά αποχές δεκτή 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή Πέτει <clears throat> 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρα 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήτρα 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 118 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 118 ηλεκτρονικός έλεγχος. Συφίσατε όλοι πέρα στι οφθαλμούς; 28, 27, 510 υπέρ. Κατά αποχής. Δεκτή. 510 υπέρ. Κατά αποχής. Δεκτή. Ενοπήμενο 8 υπέρ. Κατά αποχής. Δεκτή. 121 υπέρ κατά αποχές 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 123 υπέρ κατά αποχές δεκτή 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή 126 υπέρ κατά αποχές, έλλειψη σαφήνειας, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 126. Ψηφίσατε όλοι, όλες. Πέρας. 23-31 απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Αιτιολογικές αναφορές. 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτεί 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτεί 9 κατά αποχές δεκτή. Αιτιολογικές σκέψεις 5-5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 11 υπέρ κατά 11 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. 27 και άλλα 27. Ισοψηφία, άρα απόρριψης για την 11. 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, η 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή, τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα. Άρχεται η ψηφοφορία. Όλοι ψηφίσατε. Λείπουν τρεις ψήφοι ακόμα. Ψηφίσατε όλοι, όλες. Πέρας. 53-0. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον Ρίχαρτ Ζέμπερ στον υδάτινό μας εμπειρογνώμονα. Δεκατέσσερα, πάλι του κυρίου Ζέμπερ για insider dealing και χειραγώγηση αγοράς. 21, 23, 24 και 25 ομού. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθήσαν. 4. Υπέρ. Κατά. Για την 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές Ποιο να ξέρει. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας πληροφορίε. Εγκρίνεται. 8. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. 30, 31 και 32. Συλλήβδιν. Ψήφι υπέρ. Κατά απόχες απορρίπτονται. 9 υπέρ. <clears throat> Κατά απόχες δεκτή. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 και 35 ομού ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 <coughs> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10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 αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παραρτήματα 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογικές σκέψεις 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17. Α, 15, συγγνώμη. Συγγνώμη, 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψήφισατε όλοι πέρας 44 ψήφοι υπέρ 3 κατά 1 από εποχή Συγχαρητήρια στον Ριχάρδο Ζήντα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συγκεντρωμένη εργασία τους και πάμε τώρα στο σημείο 15 όπως ανέφερα το σημείο αυτό δεν θα γίνει και κλεισμένον των θυρών αλλά ηνιγμένων των θυρών και επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Πρόκειται για τροποποίηση τη οδηγία 2536 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναγνω... Ε, αναγνώριση επαγγελματικών προσώνων και του κανονισμού σε σχέση με την ε, διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματο πληροφόρηση για την εσωτερική αγορά. Μπερδεμένα φαίνονται αυτά, αλλά έχουν πολύ ψωμί. και καταρχήν να δώσω το λόγο στην <clears throat> Άνια Βάις Γκέρμπερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Ματίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό και συναρπαστικό το θέμα αυτό και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε αυτό με την παρουσία του κοινού. Είναι σημαντικό να κάνουμε τώρα μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων εγώ δεν έχω ακόμα συγγράψω την έκθεσή μου. Ελπίζω τον Ιούλιο θα μπορεί να δοθεί στην μετάφραση και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε προηγουμένως μία συζήτηση για τα θέματα αυτά. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εποφελούνται όχι μονάχα από την ελεύθερη κυκλοφορία αλλά και από την ελευθερία παροχής <clears throat> υπηρεσιών και από την κινητικότητα σε σχέση με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλον τούτο, αυτό το, σε αυτό το σημείο, 20 περίπου των περιπτώσεων του Solvit που έχουν να κάνουν με προβλήματα αυτού του είδους, ένα 20% των περιπτώσεων SOLVIT έχουν να κάνουν με τα θέματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Και αυτό φυσικά είναι και ένα σημείο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό η Κομισιόν έχει προτείνει την τροποποίηση αυτής της οδηγίας ώστε να εξασφαλίσει καλύτερη δράση της ενιαίας αγοράς για την ανάκαψη και την, τις θέσεις απασχόλησης και έτσι και προωθώντας και τη μεγαλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων με μια απλοποίηση και ε, επιτάχυνση των διαδικασιών θα έπρεπε λοιπόν αυτή η οδηγία να εξασφαλίσει μια αύξηση της κινητικότητας και αυτό είναι ιδιαίτερα <clears throat> σημαντικό για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ατόμων με ε, επαγγελματικά προσόντα και επίσης της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν στους νέους συνατότητες να μπορούν να μεταβούν σε μία άλλη χώρα μέλος τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστούν εκεί, για να εργαστούν εκεί η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς είναι η αρμόδια επί της ουσίας για το θέμα αυτό, αλλά εμείς είμαστε αρμόδιοι για τα θέματα υγείας <clears throat> και πρέπει να είναι πολύ σημαντική και η θέση που θα, θα θέσει η γνωμοδότησή μας για τα θέματα υγειονομικής περιθέλψης και γενικά θέματα υγείας. Εδώ υπάρχουν δύο πτυχές οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Από μια πλευρά είναι η κινητικότητα την οποία εμείς θέλουμε να προωθήσουμε αλλά επίσης και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη δυνατότητα κινητικότητας των ασθενών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν και την κινητικότητα και των παρεχόντων υπηρεσίες και των ασθενών κτλ. Η οδηγία αυτή καλύπτει 7 επαγγέλματα, κατηγορίες επαγγελμάτων που μπαίνουν σε αυτόματη διαδικασία αναγνώρισης και έξι από αυτά είναι στον τομέα της ε, υγειονομικής περίθαλψης. Είναι γιατροί, φαρμακοποιοί, ε, οι ΜΕΣ και οι ε, νοσοκόμες. Με αυτήν την ε, αυτόματη λοιπόν αναγνώριση θα, αυτή η αναγνώριση θα μπορεί να γίνει με μία διαδικασία συντονισμού η οποία ζητά ορισμένα ελάχιστα προσόντα σε σχέση με την κατάρτιση αυτών των επαγγελμάτων. Είναι τα ελάχιστα λοιπόν πρότυπα. Και τονίζεται και από την νομική υπηρεσία ότι γίνεται μια εναρμόνιση επί τη βάση ελαχίστων προσόντων. Θέλω τώρα να πάρω θέση για τα διάφορα <clears throat> επαγγέλματα. Καταρχήν για τους φαρμακοποιούς. Προβλέπετε μια διαγραφή της ρήτρα του άρθρου 120 παράγραφος 4 που λέει ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά προσόντα για τη δημιουργία νέων φαρμακείων. Επομένως δεν είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά προσόντα όταν πρόκειται για δημιουργία νέων φαρμακείων. Δηλαδή, αλλιώς πρέπει ο φαρμακοποιός να αναλάβει ένα υπάρχον φαρμακείο το οποίο υπάρχει τουλάχιστον τρία χρόνια ή να παραμείνει τρία χρόνια στην χώρα όπου θα πρέπει να εργαστεί. Η Κομισιό θεωρεί ότι αυτό είναι παραβίαση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας, αλλά είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ασφάλεια των ασθενών. Σε πολλά κράτη-μέλη ισχύει ότι υπάρχουν εθνικοί περιορισμοί σε σχέση με, τα, με τις άδειες φαρμακοποιών και υπάρχουν και περιφερειακές ε, περιοριστικές διατάξεις, αλλά δεν ισχύουν σε όλες τις χώρες. Είναι σημαντικό όμως αυτό για την επίτευξη μιας ε, ασφάλειας των ασθενών να μπορούν να υπόκεινται οι φαρμακοποιεί στα εθνικά συστήματα και να έχουν πλήρη γνώση όλων των φαρμακευτικών σκευασμάτων προτού ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους, δηλαδή να υπάρχει αυτή η ρήτρα των τριών χρόνων. Γι' αυτό αναρωτιέμαι γιατί η ρήτρα αυτή έχει διαγραφεί μετά και από την έκθεση αντικτύπου που, στην οποία προέβη η Κομισιόν και το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ένα άλλο θέμα που έχει πάλι να κάνει με τους φαρμακοποιούς είναι ότι η οδηγία προβλέπει οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να κάνουν μία άσκηση υποχρεωτικά επί έξι μήνες μετά από την θεωρητική τους κατάρτιση και εκπαίδευση σε πανεπιστήμια. Αυτό θα γίνεται σε ορισμένα κράτη με εύκαμπτο τρόπο, δηλαδή θα μπορούν να κάνουν ευέλικτα αυτή την άσκηση. Αυτό όμως δημιουργεί προβλήματα στη Σουηδία, τη Φιλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και πάλι Αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά στο τέλος των σπουδών αυτή η άσκηση και όχι ενδιαμέσως εάν χρειάζεται. Ερχόμαστε τώρα στους γιατρούς. Εδώ η οδηγία μειώνει από τα 6 χρόνια στις 5 500 ώρες σε 4 χρόνια, σε 5 χρόνια μάλλον, και 4-500 ώρες, αλλά σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της ε, ασφάλειας για την κατάρτιση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο αριθμός των ωρών, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χρόνων, για να γίνει σαφές ότι εξασφαλίζεται και η ε, ασφάλεια των ασθενών. Οδοντίατροι δεν αλλάζει τίποτα η οδηγία για το χρόνο εκπαίδευσης των 5 ετών, αλλά εδώ υπάρχει το εξή πρόβλημα. Για τους γιατρούς έχουμε συσσωρευτικά χρόνια και ώρες, για τους οδοντιάτρους όχι. Γιατί λοιπόν στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει μια τέτοια ρήτρα. Η Ένωση Ευρωπαίων Οδοντια... Οδοντιάτρων είχε ζητήσει πέραν των 5 χρόνων να είναι 5.000 ώρες η εκπαίδευση όπως συμβαίνει κατά αναλογία και για τους ιατρούς για να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα οδοντιατρικής περίθαλψης και η ασφάλεια των ασθενών. Ερχόμαστε τώρα σε ένα δύσκολο σημείο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο που είναι η νοσοκόμε και με Εδώ προβλέπεται από 10 χρόνια να πάνε στα 12 χρόνια συνολικής εκπαίδευσης. Αυτό είναι βέβαια ένα αμφιλεγόμενο σημείο. Γιατί στο σύστημα αυτόματης ε, αναγνώρισης είναι το μόνο στο οποίο αναφέρεται συγκεκριμένος αριθμός ε, ε, ετών εκπαίδευσης. Ενώ σε άλλα επαγγέλματα τίθεται ένα επίπεδο εκπαίδευσης ως προϋπόθεση για την αναγνώριση, αλλά δεν υπάρχει κανένα άλλο επάγγελμα στο οποίο μετράνε τόσο πολύ τα συνολικά χρόνια της ε, εκπαίδευσης. Είναι σαφές βέβαια ότι πρέπει να έχει τελειώσει κανείς το γυμνάσιο και το λύκειο προτού κάνει αυτή την εκπαίδευση, αλλά σε άλλα τα ε, επαγγέλματα δεν υπάρχει υποχρέωση για ένα συνολικό αριθμό ετών εκπαίδευσης. Ο στόχος ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται πίσω από αυτή την ρήτρα είναι ότι θέλει κανείς να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ποιότητα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς βελτιώνει κανείς την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχουν οι ΜΕΕΣ και οι νοσοκόμες όταν μονάχα μετράω τον αριθμό των ετών <clears throat> συνολικής εκπαίδευσης και δεν λαμβάνω καθόλου υπόψη το θέμα της ποιότητας της ε, και κατάρτισης. Σε ένα παράρτημα τώρα η οδηγία αναφέρει ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο αυτής της ε, εκπαίδευσης, αλλά είναι πεπαλαιωμένο και προκατακλυσμία αυτό το παράρτημα σε σχέση με το περιεχόμενό του και πρέπει να τροποποιηθεί. Η Κομισιόν δεν έχει κάνει ακόμα καμία πρόταση για το θέμα αυτό, αλλά έχει προβλέψει κάτι εξουσιοδότηση πράξης και αυτό ίσως σημαίνει ότι μόνο η Κομισιόν θα πρέπει να καθορίζει το περιεχόμενο των σπουδών. Εμείς ως κοινοβουλευτικοί και πιστεύω ότι εκφράζω όλους τους βουλευτές θα θέλαμε εμείς οι ίδιοι να έχουμε τη δυνατότητα να αριθμίσουμε το θέμα αυτό και επομένως δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε την οδό των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Θέλουμε να βελτιώσουμε λοιπόν την ποιότητα της εκπαίδευσης με το να μην είναι σαν μόνο κριτήριο ο αριθμό των ετών συνολική εκπαίδευση αλλά και το επίπεδο ποιότητα. Επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, παραδόσεις για την εκπαίδευση στην Ευρώπη. Είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσει κανείς τη συγκρισιμότητα στον τομέα αυτό. Υπάρχουν διαφορετικά διαστήματα διακοπών, παραδείγματος χάρη υπάρχουν διαφορετικά συστήματα για την ηλικία εισόδου στις ε, σπουδές αυτές. Υπάρχουν διαφορετικά όρια για την είσοδο στα νηπιαγωγεία στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Φιλανδία κτλ. Είναι διαφορετικά από τις άλλες χώρες και έχουμε πολλές διαφορές εν τέλει σε σχέση με τις αρμοδιότητες που έχουν οι, τα επαγγέλματα αυτά. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις αυξάνονται υποχρεώσει για την αναγνώριση, αλλά τελικά τα καθήκοντα καθορίζονται σχεδόν αποκλειστικά από τα κράτη-μέλη για αυτά τα επαγγέλματα. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να πούμε ότι έχουν αυξηθεί οι απαιτήσει, γιατί είναι διαφορετικέ οι αρμοδιότητε και υπάρχουν μεγάλε διαφορέ και στα συστήματα εκπαίδευση. Στο ψήφισμά του του Νοεμβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει ότι η λεγόμενη δυτή αναγνώριση, διπλή εκπαίδευση, διπλού είδου εκπαίδευση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και επομένω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο χρόνο εκπαίδευση ή κατάρτιση ο οποίο λαμβάνει η κάτα ο οποιου λαμβανει μέσα στα πλαίσια τη λεγόμενη διτή εκπαίδευση, δηλαδή και σε επαγγελματικού χαρακτήρου, χαρακτήρα σχολέ. Υπήρξε και μια ακρόαση στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για το σύστημα αυτό που υπάρχει σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Λουξεμβούργο ή στις κάτω χώρες και στη Γερμανία, αλλά υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν εναλλακτικά την επαγγελματική <clears throat> ε, εναλλακτική ή διαδοχική σχέση μεταξύ <clears throat> των, ε, της σχολικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ άλλα επιτρέπουν την παράλληλη ε, εκπαίδευση. Σε ορισμένα συστήματα λοιπόν η πρακτική εκπαίδευση γίνεται μονάχα στο τέλος των θεωρητικών σπουδών. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι πιο επωφελές σε σχέση με την ποιότητα. Επίσης υπάρχουν τα συστήματα αυτά της διτής ε, κατάρτισης εκπαίδευσης που έχουν μια πολύ χαμηλή ανεργία των νέων. Στην Αυστρία, παραδείγματος χάρη, είναι μονάχα 8,6 και 9,3 στις κατοχώρες, 15,1 στη Δανία και 7,9 στην Γερμανία η ανεργία των νέων. Συζητάμε πολλές φορές για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο και μέσα στα πλαίσια αυτής της συζήτησης Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι αυτή, αυτά τα συστήματα διτής ε, κατάρτισης να μπορέσουν να τύχουν μίμησης και από άλλες χώρες γιατί είχαμε μεγάλες επιτυχίες με αυτές. Εν συμπεράσματι με αυτή την αμοιβαία αναγνώριση δεν θα πρέπει να κινηθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε οι εθνικές επιτυχίες, τα επιτυχή μοντέλα τα οποία έχουν δείξει την αξία τους να χαθούν και να έχουμε μονάχα μία ε, πανεπιστημιακή μονάχα εκπαίδευση η οποία σε ορισμένε χώρες όπως στις, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δώσει αρνητικά αποτελέσματα. Βλέπουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι το ποσοστό των, ε, του νοσοκομιακού προσωπικού που δεν έχει ουσιαστικά προσόντα έχει αυξηθεί πάρα πολύ και έχει μειωθεί ε, πολύ και το ποσοστό του ειδικευμένου προσωπικού γιατί τελικά πολλοί από αυτούς προτιμούν τις διοικητικές θέσεις και όχι το να είναι ιατρικό προσωπικό. Υπάρχει μια σχετική έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο που αναφέρει ότι υπάρχει ακόμα και απάνθρωπη μεταχείριση των εργαζομένων στον τομέα αυτό και επομένως θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο παραλληλισμός των διαφόρων συστημάτων και εγώ πιστεύω ότι εάν θέλουμε να έχουμε μία εκ των, ε, εκ των κάτω προς τα κάτω εναρμόνιση, δηλαδή, θα πρέπει κάποια κράτη-μέλη το οποίο το, τα οποία το επιθυμούν να θεσπίζουν υψηλότερα κριτήρια. Εάν λοιπόν θέλουν να επιμείνουν ορισμένα κράτη να δίδουν ένα πανεπιστημιακές σπουδές, αυτό δεν πρέπει να εμποδίζει τους άλλους να ακολουθούν τα δικά τους συστήματα, πόσον μάλλον εάν έχουν αποδείξει την αξία τους. Η... Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση την οποία εγώ θα ήθελα να θέσω. Μερικά ακόμα περισσότερα σημεία στα οποία θέλω να συντομογορήσω. Προτείνεται και μια απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, πιστεύω. Επίσης πρέπει να πω ότι η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει ορισμένα χρονικά όρια, τα οποία μου φαίνονται ιδιαίτερα φιλόδοξα. Προβλέπουμε και μία μορφή ιονή αναγνώρισης. Αν ένα κράτος μέλος λοιπόν δεν κάνει εγκαίρως την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, αυτό σημαίνει ότι γίνεται μια σιωπηρή έγκριση των προϊόντων αυτών, αλλά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το προβληματικό, διότι θα πρέπει να βασιζόμαστε απόλυτα στην ποιότητα των προσόντων αυτών για λόγους υγείας και προστασίας των ε, ασθενών. Είναι επίσης να σημαντικό όταν για κάποιον δεν υπάρχει απαγόρευση συνέχισης της ε, εκπαίδευσης στον υγειονομικό τομέα, να μην μπορεί να ζητήσει εκπαίδευση σε ένα άλλο κράτο μέλο. Αυτά τα στοιχεία για την απαγόρευση θα πρέπει να στέλνονται στην Κομισιόν και επομένω υπάρχει αυτό ο μηχανισμό απαγόρευση ο οποίο προστατεύει του ασθενεί. Και άλλα δύο σημεία, τα άλλα πάρα πολύ γρήγορα. Το θέμα των γλωσσικών γνώσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδίω για τα θέματα τη ε, υγειονομική περίθαλψη είναι απαραίτητο να υπάρχουν πλήρε γλωσσικέ γνώσει. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε και το πώ γίνεται ο έλεγχο των γλωσσικών <laughs> δυνατοτήτων. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητε ενέργειε ώστε η αναγνώριση αυτή να βασίζεται στι απαραίτητε γλωσσικέ γνώσει και να μπορεί κανεί να εξασφαλίζει ότι μπορούν να γίνονται από ανεξάρτητου φορεί, όπω είναι οργανώσει ασθενών και εδώ θα, θα πρέπει να βρούμε και άλλου τρόπου ενδεχομένω για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αποτελεσματικέ γλωσσικέ γνώσει και όχι μοναχά εν μέρη και αποσπασματικέ και εμβαλωματικέ γνώσει, ώστε να μπορεί τελικά ο ασθενής να γνωρίζει ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του, του υγειονομικού προσωπικού και επομένως ότι αυτά τα προσόντα τα οποία έχει αποκομίσει κάποιος τον υγειονομικό προσωπικό μπορούν να είναι έγκυρα και σε άλλες χώρες. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά είναι σημαντικά να αντιμετωπιστούν και όλα αυτά θα προσπαθήσω να διεξέλθω στην έκθεσή μου και τέλος για την κατεξουσιοδότηση νομική πράξη και εδώ έχω αμφιβολίες, πιστεύω, ότι ιδίω σε ό,τι αφορά την, ε, το περιεχόμενο της ε, ε αυτό πρέπει να είναι θέμα του νομοθέτη και δεν μπορούμε να το αφήσουμε στα χέρια της Κομισιόν με κατεξουσιοδότηση πράξη και γι' αυτό έχω μια αντική θέση για το θέμα αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ και για την ανταλλαγή απόψεων που έχουμε κάνει με τους κοιόδης και ελπίζω ότι και μέσα στην Επιτροπή μας από την ανταλλαγή αυτών απόψεων θα έχουμε και νέα στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να ενσωματωθούν στην έκθεσή μου με τον κύριο Πρέμπολς, την κυρία Πρέμπολς και με άλλους συναδέλφους έχουμε κάνει ήδη επαφές. Θα τις κάνω και με τα, τους άλλους και συγγητές και σας ευχαριστώ τα μάλα. Ευχαριστούμε πολύ, <clears throat> Άνια, για την εισαγωγή αυτή που έκανες, για την παρουσίασή σου. Πολύ καλή. Ο Μάριο Πυρίλο πρώτα απ' όλα, σκιώδης ηγητές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο, η οποία με εξαιρετικό τρόπο περιέγραψε τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε. Είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων στο Στρασβούργο και είδαμε επί σημείο συμφωνούμε και επί όχι. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μου φαίνεται πολύ ε, ισορροπημένη. Τα καινοτόμα στοιχεία τα οποία είχαν ήδη αναδειχθεί στην πράσινη βίβλο και τώρα βρίσκονται στο νομοθετικό κείμενο, με βρίσκουν σύμφωνο ε, ε, και διότι καταφέρουν, καταφέρουν να ξεπεράσουν τα προσκόμματα της ε, κινητικότητας τα οποία έχουν αναφερθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες την δυνατότητα να επιτύχουν γρήγορη αναγνώριση των προσόντων τους και επομένως ε, θα ε, διευκολυνθεί η κινητικότητα. Το νέο άρθρο 57, αυτά του ενιαίου ΓΚΙΣΕ, θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν ε, πληροφόρηση σωστή από ένα και μόνο σημείο και θα δώσει στους ε, ετούμενους την δυνατότητα να ξεκινήσουν την διαδικασία αναγνώρισης επιγραμματικά. Αυτό που με βρίσκει επίσης σύμφωνο είναι η ε, απλούστευση και η διευκόλυνση της όλης διαδικασίας γιατί με τον τρόπο αυτό λειτουργεί καλύτερα και η κινητικότητα και γίνεται και πιο λειτουργική η ενιαία αγορά. Τα κράτη-μέλη καλούνται επίσης ε, να ξαναδούν ε, την νομοθεσία σχετικά με τα επαγγέλματα τα ε, αναγνωρισμένα επαγγέλματα τα οποία είναι ρυθμισμένα ε, στις ε, χώρες τους και ε, κυρίως να δοθεί μεγάλη προσοχή όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό. Για το νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο χαίρει άμεσης αναγνώρισης το θέμα της αναγνώρισης των προσόντων θα αποτελέσει και μια διασφάλιση των συμφερόντων των πολιτών που πλέον θα αισθάνονται πιο σίγουροι. Οι γιατροί οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν πλέον και στο εξωτερικό όταν θα έχουν ήδη δουλέψει και στην χώρα τους χωρίς ε, να έχουν πρόβλημα. Το σύστημα επαγρύπνησης επίσης ε, με βρίσκει σύμφωνο γιατί διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέραμε ε, περιλαμβάνονται ήδη όχι μονάχα στην γνωμοδότηση που είχα κάνει ως εισηγητής ε, επί της ε, τροποποίησης του, ε, της οδηγίας 2005-36 αλλά και με πιο ορθό και συμπυκνωμένο τρόπο αναφέρονται και στην έκθεση που εγκρίναμε στην Ολομέλεια. Συμφωνώ τέλος με την, επικη, την επικαιροποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων κυρίως όσον αφορώ τον νοσηλευτικό προσωπικό και τις ΕΜΕΣ και συμφωνώ και με την παρακολούθηση από το προσωπικό αυτό ειδικών σεμιναρίων. Όπως είπε και η συγγήτρια, ε, πολλοί ίσως ε, δεν συμφωνήσουν με την ε, τροποποίηση αυτή, αλλά εγώ θα συμφωνήσω. Εάν θέλουμε μία πραγματικά καλή κινητικότητα μεταξύ των χωρών, τότε θα πρέπει να, να, να μπούμε στη διαδικασία της κατάρτισης στην χώρα μου. Πρέπει να σας πω ότι το λουσελευτικό προσωπικό, ε, είτε νοσοκόμοι είτε ΜΕΣ, ακολουθούν μια ε, μεγάλη διαδικασία σπουδών που ξεκινάει από το τέλος του Λυκείου και φτάνει στο Πανεπιστήμιο. Ε, και μάλιστα εμείς ε, έχουμε 13 χρόνια εκπαίδευση ενώ στην οδηγία αναγνωρίζονται τα 12 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ξεκινάμε ήδη με μια διαφορά. Η συνάδελφος αναφέρθηκε επίσης και σε στοιχεία για την ανεργία. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε αυτά να τα ξαναδούμε λίγο, διότι η πράσινη βίβλος, όπως ε, τη γνωρίζουν και την έχουν διαβάσει οι συνάδελφοι, προβλέπει περίπου ένα εκατομμύριο θέσεων εργασίας που θα πρέπει να καλυφθούν βεβαίως από ικανούς επαγγελματίες που θα έχουν αναγνωρισμένα προσόντα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει ε, να εφαρμοστεί ε, όσο γίνεται πιο γρήγορα η οδηγία αυτή ναι, και πιστεύω ότι κάναμε ήδη ένα καλό βήμα προς τα εμπρός. Η Κομισιόν δέχτηκε και κάποιες από τις, προστάσεις, από τις προτάσεις μας. Ε, τώρα συζητάμε και για όποιες δυσκολίες έχουν παραμείνει. Θα πρέπει να τις ξεπεράσουμε και αυτές. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε διαφορετικά μέτρα και σταθμά μεταξύ των χωρών ε, μελών. Και βεβαίω αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη όλοι οι συνάδελφοι και κυρίω ε, οι συνάδελφοι από τη χώρα τη ε, εισηγητρία. Αυτά λοιπόν. Θα περιμένουμε να υποβάλει και την πραγματική έκθεση, την τελική έκθεση, επί τη οποία θα συζητήσουμε. Η συνάδελφος Φρίδα Βρύπουλη έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, την κυρία Βάισμπέργκερ. για όλα τα σημεία που εντοπίζει όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και για τη δικιά μας Επιτροπή σίγουρα, αλλά είναι και ένα περίπλοκο θέμα, γιατί η κινητικότητα των εργαζομένων όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Τώρα μάλιστα που ο πληθυσμός ε, γερνάει, έχουμε πιο πολλούς ηλικιωμένους, αλλά και επειδή η υγεία είναι ένας ε, πολύ ε, χαρακτηριστικός τομέας απασχόλησης. Γι' αυτό οι αποφάσεις που θα πάρουμε πρέπει να είναι καλές. Τόνισε και η συγγήτρια ότι η ασφάλεια του ασθενούς πρέπει να είναι το σημείο κίνησης για ό,τι απόφαση πάρουμε. Μίλησε επίσης και για μια ενδιαφέρουσα ακρόαση που Επιτροπή ΙΜΚΟ έκανε στις 25 Απριλίου. Σίγουρα εκεί ακούσαμε πάρα πολλά, μας δόθηκε πολύ τροφή για σκέψη. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα μας δίνεται ευκαιρία εδώ να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας και να ανταλλάξουμε έτσι απόψεις και να ξεκαθαρίσουμε κάποιες αμφιβολίες που υπήρχαν. Εγώ χτες για παράδειγμα νόμιζα ότι πρόκειται μόνο για τη γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής, ότι μόνο αυτό θα συζητούσαμε σήμερα. Ενώ εδώ μιλάμε για το θέμα αυτό γενικότερα. Έχω λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις για διάφορα σημεία και στο μέλλον θα τις παρουσιάσω. Τώρα, η παράταση του βασικού χρόνου σχολικής εκπαίδευσης από 10 στα 12 χρόνια που βλέπουμε στο άρθρο 31, εγώ αντιλαμβάνομαι από την πρόταση της Επιτροπής αλλά και από τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας ότι προς το παρόν 24 από τις 27 χώρες μέλη έτσι κι αλλιώς εφαρμόζουν τον κανόνα αυτό των 12 ετών. Θέλω επίσης να ρωτήσω την Επιτροπή να μου πει ποιες είναι οι τρει αυτές χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν αυτό τον κανόνα ακόμα. Και γνωρίζουμε γιατί δεν το κάνουν. Ή τι προβλήματα ε, μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ώστε να μην εφαρμόζουν τον κανόνα των 12 ετών. Πώς το εκτιμάει αυτό η Κομισιόν. Ό,τι πληροφορίες έχει αυτό να μας πει. Το δεύτερο που με ενδιαφέρει είναι στο άρθρο 4 το θέμα της ε, επαγγελματική κάρτας. Είναι κάτι που προτάθηκε και εγώ κατάλαβα ότι εκφράστηκαν πολλές ανησυχίες μια τέτοια κάρτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει όμως ποτέ μια πραγματική αναγνώριση. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις. Έπειτα το κόστος. Εδώ χρειάζεται νομίζω μια διευκρίνηση. Τρίτον, από την ακρόαση φάνηκε ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και για την μερική αναγνώριση. Είναι πολύ δύσκολο να οριστεί κάτι τέτοιο ιδίως στον τομέα της υγείας. Μια τέτοια προσωρινή αναγνώριση είναι δύσκολο και να την ορίσουμε και να την εφαρμόσουμε στην πράξη. Σίγουρα θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα στην πράξη. Έπειτα αυτή η προσωρινή αναγνώριση σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, ε, δεν μπορεί να αποτελέσει τον κανόνα. Είναι δηλαδή ένα σημείο αυτό το οποίο τους καλώς πρέπει να κοιτάξουμε παρατέρω. Τέλος, όσον αφορά τις γλωσσικές ε, γνώσεις, το αφρο 53 δηλαδή και τη λογική σκέψη 19, πρέπει οι γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό να μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή απρόσκοπτα την ιατρική πρακτική. Άρα θα πρέπει να έχουν τέτοιες ε, γνώσεις. Υπάρχει μια περίπτωση, υπόθεση Χάιμ για παράδειγμα, όπου αναφέρεται σαφώς ότι η επικοινωνία του δοντογιατρού με την ασθενή και οι διοικητικές οργανώσεις και τα λοιπά θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικές οι γλωσσικές γνώσεις. Δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας, αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι καθοριστική σημασία να μπορεί να υπάρχει η επικοινωνία στα ιατρικά επαγγέλματα. Εδώ στο Βέλγιο αναφέρεται σαφώς στην νομοθεσία ως δικαίωμα του ασθενούς να μπορεί να επικοινωνήσει δηλαδή στην ε, γλώσσα του. Σε πολλές χώρες μέλη αναμφίβολα υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχω καταλάβει, αλλά και στις κατοχώρες και στην Αυστρία οργανώνονται και εξετάσεις για να φανεί ότι ξέρει καλά αυτός που θέλει να δουλέψει εκεί τη γλώσσα. Ώστε να μπορέσει μόνο εφόσον έχει περάσει αυτές τις εξετάσεις να εξεταστεί η αίτησή του. Η συγκήτρια αναφέρθηκε και σε αυτό. Εμένα με απασχολεί πολύ λοιπόν η διατύπωση, γιατί έτσι όπως έχει τώρα ε, δεν είναι ικανοποιητική. Ελπίζω να μπορέσουμε να την κοιτάξουμε και να τη βελτιώσουμε κάπως. Έτσι συνοψίζω λοιπόν προς το παρόν τα πιο σημαντικά σημεία που έχω να αναφέρω. Από εκεί και πέρα πιστεύω και εγώ ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία και ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε κάτι πολύ καλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Φρίντα Επόμενος ο Πίτερ Λίζα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστώ και την Άνια Βάζ για το έργο της και την παρουσίασή της. Εγώ θέλω να υποστηρίξω την Άνια ιδιαίτερα. Εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος είμαστε αρμόδιοι και για τα θέματα υγείας στα κρατημέλη. Πρέπει να ενδιαφερόμαστε και για την κατάσταση της, του ιατρικού, των ιατρικών επαγγελμάτων. Και εγώ θέλω να τονίσω αυτό το οποίο Αναφέρεται και στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας ότι είναι μια εκ, για, ε, εξελαχίστων ε, εναρμόνιση. Εγώ έχω κάνει ιατρικές σπουδές, όχι φαρμακευτικές σπουδές, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο και κατά τη διάρκεια των σπουδών να κάνουμε πρακτική άσκηση και όχι μονάχα πρώτα να γίνεται η θεωρητική κατάρτιση και μετά η πρακτική. λέει ότι πρέπει να καταργηθεί το σύστημα της ε, Σουηδίας, της Φιλανδίας και της ε, Μεγάλης Βρετανίας που γίνεται άσκηση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Βέβαια υπάρχει επικουρικότητα, θα πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια της αναγνώρισης και να δούμε και τα θέματα κριτηρίων, αλλά θα ήθελα να μου εξηγήσει κανείς γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με το φιλανδικό, σουηδικό ή βρετανικό σύστημα όπου γίνεται πρακτική εξάσκηση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και όχι μονάχα στο τέλος της θεωρητικής εκπαίδευσης. Εμένα μου φαίνεται και απόλυτα λογικό κάτι Για τους ιατρούς θέλω να υποστηρίξω αυτά τα οποία ανέφερε προηγουμένως η Άνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο όταν αφαιρείται η άδεια άσκησης από ένα ιατρό ή υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει αυτή την άδεια άσκησης θα πρέπει να υπάρχει ταχεία πληροφόρηση. Γνωρίζει ο πρόεδρος το πρόβλημα που είχαμε πρόσφατα στη Γερμανία. Ένας Ολλανδός ιατρός είχε χάσει την ικανότητα να ασκεί το ιατρικό επάγγελμα. Παρ' όλα αυτά και στη δική του εκλογική περιφέρεια και στη δική μου εκλογική περιφέρεια συνέχισε να εργάζεται ως ιατρός. Και αυτό γιατί δεν υπήρξε ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών. Και σε αυτό είναι πολύ σωστή η πρόταση της Κομισιόν. Επίσης με την άνοια έχω κάποιο πρόβλημα για την ε, αυτόματη αναγνώριση η οποία μπορεί να προκύψει από την εκπνοή των προθεσμιών αναγνώρισης ότι με τον τρόπο αυτό αφήνουμε ελεύθερο στη φύση και στους ασθενείς κάποιον για το λόγο αυτό. Τώρα για τις ε, ε, νοσοκόμες τους και τις νοσοκόμες και τις ΜΕΣ και τα λοιπά. Και πάλι μιλάμε για μια ελάχιστη εναρμόνιση. Αν είναι 13 χρόνια εκπαίδευση στην Ιταλία, εντάξει, δεν μπορώ να επιβάλλω οτιδήποτε επί τη βάση μιας χώρας, το να είναι 10 ή 12 ή 13 χρόνια. Αλλά σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, υπάρχει δυνατότητα μετά από 10 χρόνια συνολικής εκπαίδευσης να μπει κανείς στο επάγγελμα του, της νοσοκόμου ή μέας. Και δεν θεωρώ ότι το να έχει κανείς ε, απολυτήριο λυκείου είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο γιατί έχω γνωρίσει πολλές μέες και νοσοκόμους που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους χωρίς να έχουν τελειώσει το λύκειο. Δεν πρέπει λοιπόν να εμποδίζεται λόγω της ε, έλλειψης απολυτηρίου να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορώ. Να φανταστώ λοιπόν ότι προκύπτει πρόβλημα με την ε, δραστηριότητα αυτών των ε, ε, νοσοκόμων και μεών επειδή δεν έχουν απολυτήριο λυτήριο. Άμα κάνουμε αυτό το, το θεωρήσουμε αυτό δεδομένο ότι πρέπει να έχουν απολυτήριο λυκείου, τότε ουσιαστικά δημιουργούμε μια άλλη τάξη ιατρικού προσωπικού που δεν έχουν καθόλου ε, πτυχίο σε επίπεδο λυκείου ή λίγο πιο κάτω και έχουμε και την εμπειρία της αγγλικής ε, έρευνας αυτής που δείχνει ότι πράγματι άμα έχουμε πολύ υψηλές απαιτήσει, τελικά είναι το ανειδίκευτο προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της περίθαλψης και αυτό αποβαίνει σε, βάθο, σε βάρος του ε, ασθενούς. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια διόρθωση της πρότασης της Κομισιόν. Θα ήθελα να ζητήσω από την Άνια Βάσκη να κάνει μια πιο συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα αυτό, ώστε να μην υποχρεωθούν τα κρατη να μειώσουν την, ε, ε, το επίπεδο εισόδου αλλά και να μην θεωρείτε ότι η ποιότητα είναι μονάχα θέμα ετών ε, εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Είναι και ο πρώτος Πέτερ Λίζερ. Έχουμε την ίδια μοίρα βέβαια και εσύ και εγώ για, για τις εκλογικές μας περιφέρειες με τον Ολλανδό αυτό ιατρό ο οποίος πέρασε τα σύνορα παρά το γεγονός του είχε απαγορευτεί η εργασία ως ιατρού στις κάτω χώρες. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να βρει τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να αποτρέψει τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα το γενικό θέμα της περίθαλψης και των ε, ιατρικών επαγγελμάτων, έχουμε την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Εγώ επειδή έρχομαι από τη Γερμανία θα ήθελα να έχω μια ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για την πρόταση Κομισιόν. Υπάρχει δυνατότητα να κάνει κανείς μια κατάρτιση χωρίς να έχει την πρόθεση να πάει σε μια άλλη χώρα μέλος. Δηλαδή να ε, είναι περιοριστικό αυτό το στοιχείο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω την άποψη της νομικής υπηρεσίας και μετά θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Από αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς, όταν, από τη στιγμή μάλλον που καλύπτονται οι απαιτήσει, βεβαίως η κατάρτιση μπορεί να λάβει χώρα στη Γερμανία ή αλλού. Γεγονός είναι ότι εάν η εναρμόνιση αφορά τα 12 χρόνια, ε, τότε η Γερμανία θα μπορεί να δώσει την, ε, ε, τα όσα αναφέρονται στο παράρτημα 5, θα μπορεί να τα εγκρίνει. Με άλλα λόγια δηλαδή, η απόδοση προσόντων του παραρτήματος 5 ε, είναι θεραπευής της ε, κάλυψης των άλλων προηγουμένων απαιτήσεων. Ε, δηλαδή 10 χρόνια γενική εκπαίδευση και μετά βεβαίως η παρούσα κατάσταση έτσι όπως ισχύει στη Γερμανία θα μπορούσε να συνεχιστεί. Εάν όμως ε, οι απαραίτητες προϋποθέσεις ε, ανεβούν στα 12 χρόνια τότε δεν θα μπορεί να δώσει την ε, αναγνώριση προσόντων στον νοσηλευτικό προσωπικό και στις ΜΕΕ στη Γερμανία σύμφωνα με το παράρτημα 5. Δεν θα μπορεί πλέον. Σας ευχαριστώ για τη διευκρίνησή σας και θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την Κομισιόν να λάβει το λόγο. Να λάβει θέση για τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Παρακαλώ. Ε, ε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να έρθουμε και να απαντήσουμε στα πάρα πολύ ενδιαφέροντα σχόλια και την συζήτηση που έχετε εδώ σχετικά με την πρότασή μας. Τέσσερα σχόλια έχω για τα όσα άκουσα. Πρώτον, αναθεώρηση των κανόνων της οδηγίας που έχει να κάνει με τα επτά επαγγέλματα στο οποία αναφέρθηκε και η συγκήτρια. Ο λόγος για τον οποίο θέλαμε να κάνουμε την ενημέρωση αυτή είναι να λάβουμε υπόψη μας τις εξελίξεις την περίοδο που πέρασε από τότε που εγκρίθηκε η οδηγία αυτή. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι χώρες μέλη, η διοίκηση κτλ. έχουν περάσει από Η πρόταση λοιπόν που βλέπετε αντικατοπτρίζει τις συζητήσεις που είχαμε με όλους αυτούς τους φορείς και προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας όλες τις εξελίξεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώς και να δούμε και τι γίνεται και επιτόπου στους χώρους εργασίας. Γι' αυτό και μερικές φορές για τους γιατρούς για παράδειγμα ζητήσαμε ή προτείνουμε να χαμηλώσει ο αριθμός των ετών αλλά ο αριθμός των ωρών να γίνει υποχρεωτικός. Σε άλλα επαγγέλματα δεν κάναμε αλλαγές. Τώρα υπήρξε ένα επάγγελμα που συζητήθηκε ιδιαίτερα σήμερα και αυτό είναι η νοσοκόμη. Γιατί εμείς προτείνουμε να αυξηθεί ο αριθμός των ετών από τα 10 στα 12. Ο λόγος είναι ότι θέλουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει που υπάρχουν βάσει της κατάστασης σε διεθνές επίπεδα. Για παράδειγμα, ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας λέει ότι ελάχιστη κατάρτιση πριν αρχίσει ένας νοσοκόμος να εκπαιδεύεται για νοσοκόμος πρέπει να είναι 12 έτη. Άλλες χώρες βέβαια είναι αλήθεια έχουν χαμηλότερη περίοδο. Η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία είναι αυτές οι τρεις χώρες. Η Αυστρία βέβαια σκέφτεται να ανεβάσει ε, τον αριθμό στα 12 χρόνια στο μέλλον. Εμείς καταλαβαίνουμε και το καταλάβαμε όταν κάναμε και την πρόταση ότι αυτό θα επηρεάσει άμεσα ή έμεσα την κατάρτιση και τα συστήματα υγείας. Και γι' αυτό και στην πρότασή μας λέμε 12 χρόνια ή αντίστοιχο ισοδύναμο. Γιατί ακριβώς έχουμε αυτή την ιδέα ότι υπάρχουν διαφορετικά συστήματα κατάρτιση στι διάφορε χώρε μέλη, υπάρχουν διαφορετικά συστήματα υγεία επίση κλπ. Και θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι η πρότασή μα δεν θα είναι άκαμπτη. Λέμε 12 χρόνια ή ισοδύναμο. Εμεί τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται συζήτηση με τι χώρε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι διάφορε επίτροπε, ότι ίσω παρερμηνευτεί αυτό ή φανεί ότι είναι δύσκολο να δεχτούμε κάτι ισοδύναμο. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί στο στάδιο αυτό να συζητήσουμε προκειμένου να καταλήξουμε σε μία αποδεκτή λύση. Λύση η οποία θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι λειτουργική και δεύτερον να είναι εφαρμόσιμη διότι αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι να δημιουργήσουμε φραγμούς εκεί όπου δεν υπάρχουν φραγμοί σήμερα. Συνεπώς, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι νοσοκόμοι καταρτίζονται με έναν τρόπο τέτοιο που να αντικατοπτρίζεται στις ανάγκες που υπάρχουν στην πράξη. Αλλά προσπαθούμε να δούμε με ποιο καλύτερο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Αυτό θα έρθει στους επόμενους μήνες, έχοντας συζητήσει με το Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε σε μια ιδιαίτερα αποδεκτή λύση. Αυτά όσον αφορά τα ειδικά επαγγέλματα. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα, στην οποία αναφερθήκατε και δίνει την αμοιβαία αναγνώριση ουσιαστικά. Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό για μας, διότι η ιδέα πίσω από την κάρτα αυτή, όπως είπε και η συγκήτρια, είναι να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση και να επιταχυνθεί. Για τις προθεσμίες υπάρχουν δύο σχόλια που πρέπει να έχετε υπόψη σας και να τα λάβετε υπόψη σας στην εκθεσή σας. Πρώτον, ότι πρέπει να δείτε τις προθεσμίες στο σύνολό τους, όλες τις προθεσμίες μαζί, γιατί μιλάμε για μια διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεύτερον, κάτι πολύ πιο σημαντικό και που δεν είναι αρκετά ορατό τώρα είναι ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα θα είναι ένα κλειστό σύστημα. Δηλαδή θα πρόκειται για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και όλες οι χώρες μέλη θα γνωρίζουν ποια είναι η αρμόδια αρχή που ασχολείται με αυτή και θα μπορούν και μεταξύ τους να επικοινωνούν με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του IMI. Άρα δεν μιλάμε για μια κατάσταση όπου διάφορες αρχές δεν θα γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν θα ξέρουν ποια είναι η αντίστοιχη αρμόδια αρχή σε κάποια άλλη χώρα, οπότε θα υπάρχουν καθυστερήσεις μπρος-πίσω για να μπορεί κανείς να ενημερωθεί. Όχι, μιλάμε για ένα κλειστό σύστημα όπου όλα τα έγγραφα, όλε οι προποθέσει θα είναι γνωστέ από την αρχή και όλε οι αρχέ θα ξέρουν ποιο είναι ο ομολογό του στις υπόλοιπε χώρε. Οι επαφέ μεταξύ των αρχών και οι επαφές με τον Τούντα ε, θα είναι πολύ συγκεκριμένες και ορισμένες από την αρχή. Οι προθεσμίες λοιπόν πρέπει έτσι να εξεταστούν για να πει κανείς κατά πόσο είναι λογικές ή όχι. Έρχομαι τώρα στην άρρητη αναγνώριση. Υπάρχει και κάτι που πρέπει να θυμηθούμε. Μιλάμε για αναγνώριση προσόντων αλλά όχι για άδεια άσκησης επαγγέλματος. Συνεπώς, μπορεί να έχετε την αναγνώριση της των επαγγελματικών σας προσόντων, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δικαιούστε ότι έχετε και άδεια για να ασκήσετε το επάγγελμα. Σε πολλές χώρες υπάρχουν επιπλέον απαιτήσει προκειμένου ένας επαγγελματίας να πάρει άδεια άσκησης επαγγέλματος και όπου ισχύει αυτό θα συνεχίσει να ισχύει. Ακόμα μάλιστα και σε περιπτώσεις όπου έχει αναγνωριστεί το επαγγελματικό προσόν, αλλά όχι έγκαιρα. Συνεπώς αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Τρίτον, για την μερική πρόσβαση, μερική αναγνώριση. Έχουμε μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επ' αυτού. Και τι προσπαθούμε να κάνουμε, να συμπεριλάβουμε αυτά που είπε το δικαστήριο, ότι είναι τρέχον δίκαιο, στην πρότασή μας προκειμένου να υπάρχει νομική βεβαιότητα για όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές και αρχές. Και είναι σημαντικό. Πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο όσο προχωράνε οι διαπραγματεύσεις. Γιατί βλέπετε ε, συνήθως μία μερική πρόσβαση θα έπρεπε να απορρέει από την εφαρμογή της πλήρους άσκησης. Αν λοιπόν η πλήρης άσκηση δεν είναι δυνατή, τότε συνεχίζει την μερική πρόσβαση το κράτο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κάποιο επαγγελματία να πάει και να ζητήσει μερική πρόσβαση. Όχι. Θα είναι το τέλο της διαδικασία εφόσον δεν δοθεί η πλήρη πρόσβαση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Και εσείς να το ξέρετε όσο προχωράτε με την έκθεσή σας αυτό. Τέταρτο θέμα. Οι γλωσσικές εξετάσεις. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Κατά τη γνώμη μας, είναι ήδη ξεκάθαρο με την ε, τρέχουσα οδηγία. Εκεί που λέει η οδηγία ότι ο επαγγελματία πρέπει να έχει τα γλωσσικά προσόντα προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, άρα όχι οποιασδήποτε γλωσσικέ ε, ικανότητε, λέει η οδηγία να είναι οι γλωσσικέ του γνώσει τέτοιε που να μπορεί να αποκριθεί στο επάγγελμά του, στην άσκηση του επαγγελματό του. Αυτό υπάρχει ήδη στην οδηγία. Συνεπώ, αν έχετε την υποχρέωση αυτή, ε, άρρητα κάποιο πρέπει να το ελέγχει κατά πόσο όντω έχετε τι γλωσσικέ αυτέ γνώσει ή όχι. Με την πρότασή μα θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε να γίνει αυτό σαφές και να προτείνουμε ίσως και κάποια βήματα ώστε να δούμε πώς οι διοικήσει, οι αρχές θα μπορέσουν να προχωρήσουμε αυτή την απέτηση. Θα συζητηθεί παρατέρο βέβαια και ελπίζουμε ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε έναν καλό συμβιβασμό. Όμως, κάτι που θέλω να τονίσω είναι τι θέλουμε να αποφύγουμε. Να μην γίνονται δύο φορές αυτές οι εξετάσεις. Μην φτάσουμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου ένας επαγγελματίας ζητάει πρόσβαση για να μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμα σε μια άλλη χώρα. Ε, δίνει εξετάσεις στις αρχές και μετά ξαναδίνει εξετάσεις και για τον εργοδότη. Δηλαδή δύο φορές κάνει το ίδιο πράγμα. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Γι' αυτό και λέμε οι γλωσσικές εξετάσεις δεν πρέπει να αποτελούν μέρο της διαδικασία αναγνώρισης, αλλά πριν του δοθεί η άδεια άσκηση επαγγελματο. Και το δεύτερο είναι ότι μία φορά πρέπει να δίνουν τέτοιε γλωσσικέ εξετάσει. Αυτά είχα να πω προς το παρόν. Κάτι τελευταίο μόνο. Είμαστε ανοιχτοί και διαθέσιμοι να συζητήσουμε με την Επιτροπή σας και με όλους τους ευρωβουλευτές και διμερώς για όλα τα θέματα που σας απασχολούν. Γιατί βλέπετε στο τέλος το τελικό προϊόν της διαδικασίας αυτής πρέπει να είναι κάτι που να είναι πολύ χρήσιμο για τους πολίτες μας και τις αρχές των χωρών μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις που δώσατε και τις ε, Εξήγησης. Πρωτού δώσω το λόγο στην ε, εισηγήτρια. Θέλω να χαιρετήσω μια ομάδα καλεσμένων που τους έχει φέρει ο Μάριο Πυρίλο από την Καλαβρία. Είστε ρε. Η Άνια, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πολύ καλή συζήτηση. Μπορώ να πω συνοπτικά ότι η πρόταση της Κομισιόν έχει πολλά θετικά στοιχεία και μπορώ να την υποστηρίξω και ελπίζω ότι μαζί με την Κομισιόν θα μπορέσουμε να διευθυνήσουμε καλύτερα τα σημεία αυτά. Εν πάση περιπτώσει ο μηχανισμός αυτός μου φαίνεται ότι είναι θετικός και ο μηχανισμός για την, ε, τα γλωσσικά τεστ πρέπει να λειτουργήσει σωστά και επίσης για τη μερική πρόσβαση θα πρέπει να το δούμε καλύτερα στον τομέα αυτό και για το θέμα των ελαχίστων προδιαγραφών για τις, ε, για τις νοσοκόμους. Το να έχουμε 10 χρόνια σε μια χώρα σαν όριο, αυτό δεν σημαίνει πρέπει οι άλλες χώρες να κατεβάσουν τα δικά τους ε, όρια, αλλά αν πηγαίνουμε στα 12 χρόνια γενικά, θα πρέπει οι χώρες οι οποίες έχουν ένα σύστημα διπλής κατάρτισης με πρόσβαση στα 10 χρόνια. Αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει το σύστημα αυτό της διπλής εκπαίδευσης να μπορεί να μεταλαμπαδευτεί και αλλού. Δεν πρέπει τελικά λοιπόν αυτό το σύστημα να οδηγήσει σε περιστολή της ε, κινητικότητος λόγω παραδείγματος του χρόνου ε, εκπαίδευσης και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό που έκανε η Κομισιόν η οποία έχει βασιστεί σε ισοδύναμα εκπαίδευση και πιστεύω λοιπόν ότι το να έχουμε τη διατήρηση των συστημάτων και να κρατήσει το καθένα το δικό του, εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα της Κομισιόν, λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο ε, που έχει να κάνει με την πρόταση τη Κομισιόν. Θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο, όπω και με την κυρία Μπρέπουλ, γιατί απαιτείται ένα ορισμένο αριθμό ετών κατάρτιση πριν ξεκινήσει η εκπαίδευση. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη διευκρίνηση για όλα αυτά τα σημεία και αυτό θα βελτιώσει την πρότασή μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρο, κύριε Βάι Γκέρμπερ για τα τελικά σα σχόλια και στις 8 Δεκεμβρίου Σεπτεμβρίου, μάλλον όχι Δεκεμβρίου, θα κάνουμε συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας Περιβάλλοντος με το σχέδιο της γνωμοδότησης. 20 Σεπτεμβρίου θα είναι η υποθεσμία για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 10 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία στην Αρμόδια Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου αυτό είναι λοιπόν το στενό χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι χθερινέ διακοπές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την υγεία, με την ε, περίθαλψη και τη διατήρηση των καλύτερων ε, πρότυπων σε όλα τα κράτη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ όλου αυτού οι οποίοι έλαβαν μέρο στη συζήτηση και η επόμενη συνεδρίασή μα είναι στις 20 και 21 Ιουνίου εδώ στις Βρυξέλλες. Καλή όρεξη λοιπόν και θα τα πούμε στο θερινό ηλιοστάσιο.